αλλά και στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Αυτό είναι. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Ευρωβουλευτά. Και ευχαριστώ επίση και για όλε τι παρεμβάσει Και έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το σημείο στη συζήτηση. Αύριο στις 12 η ώρα θα διεξαχθεί ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια με την ημερήσια διάταξή μας. Περνάμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη και πρόκειται εδώ για ερωτήσεις, προφορικές ερωτήσεις για απάντηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου από ετούντες άσυλο στα κράτη-μέλη και κόστος της εξέτασης των αιτήσεων αυτών των ετούντων άσυλο. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους συντάκτες αμέσως. Καταρχήν, Νάντια Χίερς. Δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνήσαμε το 2012 να έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για τη χορήγηση ασύλου αλλά σε συνδυασμό ότι παρόμοιες προϋποθέσεις και όροι θα συντρέχουν και στα κράτη-μέλη. Όμως η υλοποίηση ασυναντά αντιστάσεις και αυτό λόγω του ότι στη διαβούλευση του πακέτου για το άσυλο δεν υπάρχουν πληροφορίες, πλήρεις πληροφορίες, ανεπαρκείς πληροφορίες ή και κιόλας διαφορετικές πληροφορίες και το ίδιο συμβαίνει και για την αξιολόγηση των χρηματικών αναγκών ε, για την υλοποίηση αυτή τη οδηγία σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Πολύ λίγε πληροφορίε έχουμε. Στόχο μα λοιπόν είναι εδώ να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει μία μελέτη και να διαβιβάσει αυτέ τι πληροφορίε προ το Ευρωκοινοβούλιο. Κυρίως είναι θέματα όπω οι υπηρεσίε διαρμηνία, όπω επίση και οι υπηρεσίε ε, νομικών συμβούλων και συμβουλών που θα παρέχονται. Και δεν είναι σαφέ ποιο θα είναι το κόστο. Στην άλλη πλευρά για την αναθεώρηση των διαδικασιών αυτής της οδηγίας θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια ποιοτικά αναβαθμισμένη διαδικασία που θα είναι εποφελής για αμφότερες τις πλευρές. Θα οδηγούμαστε σε λήψη ταχαίως αποφάσεων επί αυτών των ε, αιτήσεων ασύλου ώστε να μην χρονο, χρονοτριβούμε. Και στόχος μας είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηριχθεί σε αυτό το εγχείρημα. Χρειάζονται όμως επιχειρήματα στη συζήτηση με τα κράτη-μέλη που θα δώσουν τη δυνατότητα να δούμε ποιες επιπτώσεις θα έχει η αναθεώρηση ακριβώς αυτού του πακέτου μέτρων για το άσυλο. Ιδιαίτερα η διαδικαστική πλευρά, η οδηγία όσον αφορά τις διεργασίες και διαδικασίες. Ζητούμε υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε το 2012 το πακέτο μέτρων για το άσυλο να γίνει πραγματικότητα και να καταλήξουμε σε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα χωρί ασύλου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, στη συνέχεια, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην Μόνικα Χολμάια. είναι μία από τις συντάκτριες ε, και η κυρία Χόλμαϊρ. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με τα προβλήματα της μετανάστευσης ε, και της χορήγησης ασύλου. Έχει υποβάλει αντίστοιχε προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει επακριβής ανάλυση για την υλοποίηση των υφιστάμενων νομικών διατάξεων και δεν υπάρχουν ε, και συγκεκριμένες αναλύσεις και υπολογισμοί ποιο θα είναι το συνολικό κόστος. Το ανεπιφύλακτα είναι υπέρ της προστασίας και συνδρομής εκείνων που χρειάζονται υποστήριξη και τον των τον άσυλο. Και πρέπει το δικαίωμα για χωρίση άσυλου να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη και να είναι σεβαστό, όχι όμως σε σχέση με εκείνους που θέλουν να κάνουν κατάχρηση αυτού του δικαιώματος. Και για τα 27 κράτη-μέλη πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε το οργανωμένο εμπόριο ανθρώπων να μην μπορέσει να αποκομίσει ωφέλη και να αντιμετωπίσει οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να εφαρμοστούν. Θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση για αυτούς τους ανθρώπους ότι θα βρουν προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό προβλέπονται ειδικέ διαδικασίες από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως υπηρεσίες διερμηνίας, περίθαλψη, ιδιαίτερα περίθαλψη των ευάλωτων ατόμων. Θέλω να αναφέρω κάποια σημεία τα οποία είναι προβληματικά θεωρώ. Οι αρχέ των κρατών μελών έχουν πολύ λίγε δυνατότητε να αποτρέψουν καταχρήσεις και οι επιταχυμένες συνοπτικές διαδικασίες ε, που είναι καταχρηστικές θα πρέπει να περιοριστούν. Και όταν υπάρχει παραβίαση κάποιων δικαιωμάτων ε, δεν υπάρχει δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. Και όταν ε, κάποιος επανεμφανίζεται θα πρέπει να υπάρχει μια διευρυμένη δυνατότητα μέτρων που θα μπορούσαν να ασκηθούν σε σχέση με τέτοια άτομα. Και να δούμε και την δυνατότητα επιταχυμένων τέτοιων συνοπτικών διαδικασιών μετά από την το, δεύτερο υποτροπιασμό. Αυτό σημαίνει αυξημένο κόστος. Αυξημένο κόστος και σε σχέση με τη διάθεση ε, συμβούλων, νομικών συμβούλων ή δικηγόρων που θα επικουρούν αυτούς τους ανθρώπους. Παρακαλώ λοιπόν απλά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπολογίσει τις επιπτώσεις αυτών των προτάσεών της στην καθημερινή ζωή και να δει ποιο θα είναι το διοικητικό βάρος για τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να έχουμε αναβαθμισμένο επίπεδο υπηρεσιών και δράσης, αλλά δεν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη επιβάρυνση στα κράτη-μέλη που είναι ήδη επιβαρημένα. Ευχαριστώ. Σίλβη. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ακούσουμε τη ε, λίγη γιόμ. Και η κυρία αυτή είναι συντάκτρια. Έχετε τρία λεπτά να στην παρέμβαση. Euh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι και εγώ τη συζητήσεω είναι τουλάχιστον δημιουργεί ενό καθεστώ ευρωπαϊκού ασύλου το ε, του 2012 που επιτρέπει επιτέλου να βγούμε από τι κακέ εθνικέ πρακτικέ όσον αφορά το άσυλο. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε, γιατί μα υποχρεώσει να πηγαίνουμε προ μεγαλύτερη εναρμόνιση που θα βασίζεται σε κοινού κανόνε. Είμαι πεπισμένη ότι μόνο η πρακτική συνεργασία από μόνη τη δεν θα λύσει τι αποκλήσει των εθνικών ε, συστημάτων. Θα ήθελα να πω ότι έχω ανησυχίε όσον αφορά την πρόθεση του ευρωπαϊκού συστήματο ασύλου, διότι υπάρχουν πολλά μπλοκαρίσματα σε επίπεδο ε, συμβουλίου. Τι θα γίνει λοιπόν όσον αφορά το εγχείρημα αυτό το περίπλοκο. Ε, λοιπόν, ε, τι θα προτείνει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάσωση με αναθεωρημένη πρόταση για τις οδηγίες. Ε, λοιπόν, αυτό επιβάλλεται ξαφνικά διωτική μας οδηγία αυτή η συζήτηση. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε τα αναγκαία διαδικαστικά εχέγγυα, οικονομικό βάρος να το επομιστούν τα κράτη-μέλη, το οποίο θα αυξηθεί σημαντικά για την εξέταση του ασύλου. Και τώρα περνάμε και την κρίση και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι διαδικασίες που δεν χρησιμοποιούνται καλά και αυτή η κακή ποιότητα κοστίζει στα κράτη-μέλη. Δηλαδή χρειαζόμαστε βελτίωση των ενδεικτικών ε, των πρωτοδίκων διαδικασιών που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά επιτρέψει μεσοπρόθεσμα να πραγματοποιηθούν πραγματικές εξοικονομήσεις ε, κλίμακας. Γιατί, Γιατί αυτοί οι ενορισμένοι διαδικασίες θα συμβάλλουν εξ αρχής σε καλύτερο εντοπισμό των αιτημάτων των καταχρηστικών από τις πλευράς των αρμοδίων φορέων. Και θα πρέπει να αιτιολογούνται οι αποφάσει και θα πρέπει να λαμβάνονται πιο γρήγορα οι αποφάσει που θα είναι καλύτερε ποιότητε. Άρα μείωση χρόνου διαδικασία ε, των προσφυγών, αριθμού προσφυγών και προσφυγή σε δευτεροβάθμια εξέταση κλπ. Και στο τέλο, μια γενικότερη μείωση και του κόστου. Εάν θέλουμε να αναφερθούμε στο θέμα των διαπανών, γιατί να αναφέρουμε επίση και το σύστημα του Δουβλίνου Eurodac. Γιατί κανένα κάτω μέλο δεν ζητά μία έκθεση κόστου αποτελεσματικότητα όσον αφορά την εφαρμογή του λόγου συστήματο. Ξέρουμε όμω ότι οι ανθρωπιστικέ συνέπειε είναι αξιοθρύνητε ε, και κάτι πρέπει να γίνει όσον αφορά την μεταφορά και την πρόληψη δευτερο... των άλλων μετακινήσεων στη δευτερομάθημα φάση. Λοιπόν, αν θέλουμε να μιλήσουμε για κόστος, ας το κάνουμε. Και για όλο το σύστημα, συμπραγμανούν και του κόστου του καθεστώτος του Δουβλίνου. Από την πλευρά μου, συζητείται όσον αφορά την οδηγία για τη διαδικασία, παραμένω πεπισμένη ότι το επίπεδο εναρμόνιση είναι ανεπαρκέ τώρα και ότι παρεμποδίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα τη διαδικασία. Αυτό επιβαρύνει και τα κράτη-μέλη και τα θύματα τη δίωξη το 2012 είναι στόχος μας και για λόγους σεβασμού των προθεσμιών δεν θα πρέπει να επομιστούμε την ευθύνη να καταλήξουμε σε ένα κείμενο κατακαιρματισμένο το οποίο ε, θα καταλήγει στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Θέλουμε σωστές διαδικασίες, προσβάσιμες, αποτελεσματικές. Και αυτό είναι δικός μου στόχος και αυτός της πολιτικής μου ομάδας αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντε Γιόγκ. Α, ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρο, Ε, πέρασα μια γραμμή. Η κυρία Ελέν Φλότχο είναι εκείνη η οποία θα πάρει το λόγο. Για δύο λεπτά. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, πιστεύω ότι... Δουλεύει, ε. Εντάξει. Πιστεύω ότι ο στόχο αυτή τη συζητήσεω ε, είναι να υποχρεώσουμε το Συμβούλιο να, να αποκαλυφθεί διότι έχουμε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων για το άσυλο και είναι τόσο φιλόδοξο και θα έλεγα και τόσο αναγκαίο και από το Συμβούλιο δεν έχουμε παρά μόνο ε, κάποιες, ε, κάποια εμπόδια που εμφανίζει το Συμβούλιο όσον αφορά την πρόοδο έναντι των προτάσεων που είναι επιτάπητος εδώ και καιρό. Κατανοούμε αόριστα ότι το Συμβούλιο ή τα κράτη-μέλη τέλο πάντων επικαλούνται το κόστος, αλλά όμως θα πρέπει να συνεννοηθούμε τι εννοούν. Μιλάμε ανθρώπινο κόστος, πολιτικό κόστος, οικονομικό κόστος. Και καμιά φορά αυτέ αυτές οι δαπάνες είναι αλληλένδετες. Υπάρχει και κάτι που είναι σίγουρο. Είναι οι πρακτικές που ακολουθούνται. Υπάρχει μια προστασία ελλειπή στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν δέχεται όλη τη μιζέρια του κόσμου. Το 2007, παραδείγματος χάρη, η Ευρώπη δεν δέχτηκε παρά μόνο 14% από τους πρόσφυγες του πλανήτη και ακολουθούνται πρακτικές ε, που είναι απαράδεκτες όπως στην, ε, στην Ευρώπη. Στην οι δοκιμές που γίνονται, τα τεστ και διάφορες περιπτώσεις επαναπροώθησης ε, λόγω προσφυγών που δεν έχουν αστατικό χαρακτήρα. Λοιπόν, μπορούμε να μιλούμε για κόστο, μπορούμε να μιλούμε για τι απελάσει των μεταναστών, που είναι κάτι που κοστίζει πάρα πολύ. 20.000 ευρώ κατά άτομο που απελάβνεται, λέει η Γαλλική Γερουσία. Και μπορούμε να μιλήσουμε και για το πώ μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Σίγουρα, όταν περίπου 50% των αποφάσεων πρωτόδικα ακυρώνονται στην κατόπιν εφέσεω, θα πρέπει να διαρωτηθούμε. Και αυτό κάνει η κυρία Γκυγιόμ στην έκθεσή τη, πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα τη λήψη απόφαση σε βάθμια φάση. Και έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε και κατάσταση του κόστου, του πολιτικού, του οικονομικού και του ανθρώπινου. Οι κακέ εφαρμογέ του Δουβλίνου μπορεί να επανέλθουμε πάνω σε αυτό και πρέπει να επιληφθεί το θέμα το σοβαρά το Συμβούλιο διότι και εδώ το ανθρώπινο κόστος και το οικονομικό κόστος είναι πολύ μεγάλο και το που κοστίζει πάρα πολύ κρυβά και το λένε μελέτες του Κοινοβουλίου είναι οι κρατήσεις. Οι κρατήσεις των ετούντων άσυλο έχουν απαγορευτικό κόστος. Πρέπει να το πούμε και πρέπει να το πούμε, να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε στο Συμβούλιο, είναι κατεπήγον το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Ντεγιόνγκ και αυτό συντάκτη τη ερώτηση. Έχετε δύο λεπτά, κύριε Ντεγιόν. Ευχαριστώ πολύ. Καμιά φορά είμαστε θύματα τη μεθοδολογία μα και τη δουλειά μα. Το να είχαμε μία οδηγία σε σχέση με τα κριτήρια και μία, ένα πλαίσιο για την εισδοχή θα είχαμε ε, και εδώ έχουμε μία εναλλακτική λύση ή θα αλλάξουμε αυτήν την οδηγία ή θα την εγκρίνουμε ως έχει. Αυτό θα ήταν όφελος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να το πούμε ευθύ εξ αρχής. Δεν υπάρχει, δεν θα υπήρχε ένα κοινό τέτοιο πλαίσιο χωρίς ασύλου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε όμως διαφορετικές οδηγίες και το Συμβούλιο μπορεί να ε, επιλέξει κάποιες ε, και κάποιες άλλες να τις θέσει σε ένα υποδέστερο επίπεδο. Ίσως θα μπορούσε μια νέα οδηγία Δουβλίνου να υποβληθεί, αλλά όχι μια νέα οδηγία διαδικασιών. Αυτό τι σημαίνει με άλλα λόγια. Ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν την ευθύνη για την ε, εξέταση όλων αυτών των αιτήσεων ασύλου και δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν εχέγγυα ότι σωστά θα εξετάζουν και θα αντιμετωπίζονται αυτές οι αιτήσει και σωστά θα αντιμετωπίζονται οι αιτούντε άσυλο. Γι' αυτό η ερώτησή μου πώς θα μεριμνήσετε η οδηγία αυτή να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω απώλειες και να οδηγηθούμε σε αυτής της οδηγίας. Θα προσπαθήσετε να στείλετε ένα σαφές μήνυμα των εκπροσώπων, των ερετών εκπροσώπων των πολιτών προς τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν ή θα υπάρξει προσέγγιση à la carte κατά το δοκούν από τα κράτη-μέλη που θα είναι στη δική τους διακριτική ευχέρεια. Θα πρέπει να δούμε και το κόστος. Όχι επειδή ίσως νομίζω ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι ανθρώπινα θα αντιμετωπίζονται οι τούδες άσυλο. Χρειαζόμαστε θετικέ διαδικασίες για την σωστή αντιμετώπιση τους, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ θα πρέπει να τεθεί στο πλευρό μας για να υλοποιηθούν αυτά. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και μετά από τους συντάκτες θα ήθελα να ζητήσω, να χαιρετήσω την κυρία Νίκ και που ε, βρισκόταν εδώ ο συνάδελφός μας ε, μέχρι πριν από λίγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα εξ ονόματος του Συμβουλίου την καλό να λάβει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου προσφέρετε για αυτή τη διαδικαστική οδηγία ε, όσον αφορά τα θέματα ασύλου. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα που εμπλέκονται εδώ. Οκτώ ερωτήσεις ε, στράφηκαν, απευθύνθηκαν προς το Συμβούλιο και πρόκειται πάντα για την μία και ίδια αυτή ενιαία οδηγία για διαδικαστικά θέματα και πώς θα την αντιμετωπίσουμε είναι σημαντικό λοιπόν να συζητήσουμε αυτά τα θέματα μεταξύ μας. Αναφέρεστε στην ερώτησή σας και στην έκθεση του Σεπτεμβρίου 2010, μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, πρόκειται και για την ε, έκθεση ακριβώς ε, που αφορά την εφαρμογή και υλοποίηση όλων αυτών των μέτρων από πλευρά των κρατών μελών. Αναφερόταν τότε σε αυτήν την έκθεση ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν τα αναγκαία ηχέγγυα για τις διεργασίε αυτές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να, να προαχθεί από εμάς. Να έχουμε κοινού στόχους που θα επιτύχουμε, διότι αν δεν υπάρχουν κοινοί στόχοι που θα επιτευχθούν δεν θα υπάρξει ποτέ ένα ευρωπαϊκό κοινό ενιαίο σύστημα. Τον Οκτώβριο το Συμβούλιο υιοθέτησε μία απόφαση για μία κοινή πολιτική για το άσυλο. Υπό το πρίσμα ότι δεσμεύονται τα κράτη-μέλη για τα θέματα ασύλου και μετανάστευσης από κοινού να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και θα προσπαθήσουν με συναφή, ε, συνεκτικό τρόπο να προχωρήσουν από κοινού όλα τα κράτη-μέλη με, αναμεταξύ τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε σχέση με, αυτό το, με αυτή τη συμφωνία. Ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για το άσυλο θα θεσπιστεί, θα συγκροτηθεί. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα βέβαια γι' αυτό. Γι' αυτό ζήτησε το Συμβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές τις κοινέ διατάξεις ε, να τις προτείνει, να τις εκπονήσει, ώστε να έχουμε ένα κοινό, κοινοτικό ευρωπαϊκό σύστημα για το άσυλο. Έχουμε και το πρόγραμμα της Στοχόλμης που εμπεριέχει και λέει ότι ένα τέτοιο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για το άσυλο θα πρέπει να προβλέπει την μέγιστη, τον μέγιστο εναρμονισμό που είναι εφικτός. Χρειάζεται ένα, ένας εναρμονισμός σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα επιτευχθεί. Και αυτή την όθηση την εκμεταλλευτήκαμε, αυτή την όθηση που δημιουργήθηκε και υπήρξε και υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάφορες προτάσεις. Το επισημάνατε αυτό. Αναφέρατε από πλευρά σας την Eurodac, Eurodac, αλλά ακόμα και άλλα σημεία αντίστοιχων πρωτοβουλειών, καθώς επίσης και την αλλαγή συγκεκριμένων κριτηρίων που θα πρέπει να αλλάξουν στην νέα διατύπωση, στην αναδιατύπωση αυτής της οδηγίας. Και μετά όσον αφορά επίσης και τη στέγαση, την ε, υποδοχή αυτών των ετούντων άσυλο. Και πάλι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, έχουν εκπονηθεί και έχουν διατυπωθεί σχετικές προτάσεις. Αμέσως ε, στράφηκε το Συμβούλιο και αποδίθηκε στην εργασία αυτή συγκεκριμένα και εξειδικευμένα. Εξέτασε πρώτα όλες αυτές τις προτάσεις σε βάθος, με προσοχή. Μέχρι στιγμής ε, τι συνέβαινε. Συμβαίνει μέχρι στιγμής το ότι μόνο ένας κανονισμός ε, μπόρεσε να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί σχετικά. Και πέρυσι 2010 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν πραγματικά να υπάρξει μια σε ευρύτερα πλαίσια αλλαγή αυτών των ε, διατάξεων και διαδικασιών και αυτό θα είναι υποφελές για την περαιτέρω ευδοκίμηση ενός ευρωπαϊκού κοινού συστήματος για το άσυλο. Τώρα δυστυχώς συμβαίνει το εξή Σε άλλους τομείς δεν σημειώθηκαν ε, τέτοιες πρόοδοι. Το θέμα είναι πάρα πολύ ακαθόδες και πολιτικά πολύ ευαίσθητο ευαίσθητο και γι' αυτό δεν κατέστη εφικτό μέχρι σήμερα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία επ' αυτών των πτυχών. Αυτές οι δυσκολίες πιστεύω δεν υπάρχουν μόνο σε σχέση με το Συμβούλιο αλλά υφίστανται και στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα για τις ερωτήσεις που διατυπώσατε και ε, απευθύνατε προς το Συμβούλιο θα ήθελα να αναφέρω τα εξή: Στην αναδιατύπωση αυτής της οδηγίας ε, για τα διαδικαστικά θέματα υπάρχουν αρκετά προβληματικά ζητήματα και το Κοινοβούλιο έχει ενημερωθεί επίσης, ενημερώνεται για το έργο το οποίο έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα. Και είναι απόλυτα σαφέ φυσικά ότι υπάρχουν διάφορε επιφυλάξει και, και ε, θα έλεγα αντιστάσει από πλευρά του Συμβουλίου με την νέα αυτή αναδιατύπωση αυτών των προτάσεων. Διερωτώνται οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου ποιε θα είναι οι επιπτώσει στα εθνικά συστήματα για το άσυλο. Πώ μπορεί να διασφαλιστεί ότι αυτέ οι διεργασίε θα είναι αποτελεσματικέ. Διότι αυτό είναι αυτό το οποίο επιθυμούμε. Αποτελεσματικές διεργασίε και διαδικασίε που δεν είναι δαπανηρές. Κάποια κράτη-μέλη ήταν κατά του εναρμονισμού αυτού του συστήματος μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Είπαν ότι χρειάζονται μεν κάποιε συγκεκριμένε ρήτρε και διατάξεις που θα είναι κοινέ, θα είναι κοινοτικέ και χρειάζονται και κάποια κριτήρια για την προστασία που θα είναι και αυτά κοινοτικά. Όμως το Συμβούλιο έλαβε αυτά τα πράγματα υπόψη και θα πρέπει να συνεξεταστούν. Τώρα η δουλειά είναι στα χέρια του Συμβουλίου. Είναι δύσκολο και ακαθόδες το θέμα. Βρισκόμαστε και σε μια κρίσιμη ε, οικονομική κατάσταση. Πρέπει να δείξουμε και την αλληλεγγύη μας που θα εκφράσουμε και να εκπονήσουμε προτάσεις με τις διατάξεις αυτές που δεν θα προκαλούν, δεν θα δημιουργούν υπερβολικό, καταχρηστικό, ε, ε, διοικητικό βάρος από πλευράς δαπανών. Μέχρι στιγμής δεν κατέστη εφικτό να επιτευχθεί μια τέτοια ισορροπία όσον αφορά τέτοιες προτάσεις και να αποφευθεί ότι θα υπάρξει κατάχρηση με την εφαρμογή αυτών των ε, ρητρών για το άσυλο. Και τέτοιου είδους ε, δαπανηρές καταστάσεις είναι προβληματικές για τα κράτη-μέλη. Είναι επίσης προβληματικές και για εκείνους που έχουν δικαίωμα προστασίας ε, σε διεθνές επίπεδο ως ετούντες άσυλο. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε την ενασχόλησή μας με το θέμα και να ε, μας απασχολήσει μέχρι ότου καταφέρουμε να προχωρήσουμε. Πιστεύω όμως ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα και θα τοποθετηθεί σχετικά. Είναι σημαντικό να δοθεί νέα όθηση σε αυτή τη συζήτηση νέα όθηση στο Συμβούλιο και έτσι να μπορέσει η άποψη του Συμβουλίου να ε, συγκεραστεί, να συνδυαστεί και με την άποψη της απόψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα εκφραστούν. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο στο εγγύς μέλλον. Και πιστεύω ότι, σημαντικά είναι ένα πολύ, ε, ε, ότι συνολικά είναι ένα πολύ σημαντικό πακέτο μέτρων αυτό. Μια δέσμη μέτρων με ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Όμως και τα κράτη-μέλη ρητά τοποθετήθηκαν. Είπαν θέλουν να, να, να ασχοληθούν ότι τη νέα πρόταση που θα υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακόπτεται η παρέμβαση. Ίσως όμως να αναφέρω και μια άλλη πτυχή. Συνεχίζεται η παρέμβαση. Να αναφέρω και μια άλλη πτυχή. Όσον αφορά το θέμα των δαπανών ή του κόστους ή την εκτίμηση αυτού του κόστους, αυτά τα κόστη πρέπει φυσικά να εκτιμηθούν να αξιολογηθούν. Θα συνεχίσουμε φυσικά μετά από αυτό τις διαβουλεύσεις μας στο Συμβούλιο, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε σωστά και αξιόπιστα. Για να εκτιμήσουμε σωστά και αξιόπιστα πρέπει να έχουμε πληροφορίες στα χέρια μας. Για να αποφασίσουμε χρειαζόμαστε πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει προθυμία να διαβιβαστούν, να, δια, να διαχειριστούν αυτά τα στοιχεία και να γίνουν αυτές οι αξιολογήσεις, αλλά προτού γίνει οποιαδήποτε εκτίμηση ή αξιολόγηση πρέπει να υπάρχουν οι πληροφορίες, τα πληροφοριακά στοιχεία Καλούνται λοιπόν όλοι και είναι όλοι υποχρεωμένοι να υποβάλουν, να ε, μας διαβιβάσουν τις ε, αναγκαίες αυτές πληροφορίες. Και το Συμβούλιο θεωρεί ότι αυτό το θέμα της ε, ατροποποίησης ή της αναδιατύπωσης της οδηγίας είναι πολύ σημαντικό και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και περνάει από το χέρι μας. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας και βασιζόμαστε και στηριζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το εγχείρημα. Έχει μεγάλη πραγματογνωμοσύνη, εμπεριστατωμένη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένα πλαίσιο θετική καλή συνεργασία θα μα δώσει τη δυνατότητα να σημειώσουμε πρόοδο. Πρέπει όμω ταυτόχρονα να γνωρίζουμε ότι ο στόχο ε, στόχος της, Ευρωπαϊ... της Ουγγρικής Προεδρίας είναι να καταφέρουμε σύντομα να καταλήξουμε σε ένα ευρωπαϊκό κοινό σύστημα για το άσυλο. Αυτό σχεδιάζουμε να επιτύχουμε το 2012. Θέλουμε να σημειώσουμε Θέλουμε πρόοδο από πλευρά τη Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου. Θέλουμε πρόοδο να σημειωθεί στο πολιτικό επίπεδο, αναβάθμιση να επιτευχθεί για τις ρήτρες και διατάξεις και θέλουμε πριν από το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας να έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε αυτό το ε, έργο, το εγχείρημα που έχουμε επομιστεί. Θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε καλύτερα μέσα σε ένα αρμονικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Υφυπουργέ και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Φίλε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μπορέσει να παρέμβει για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Uh, uh, ευχαριστώ. Uh, Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αυτή η οδηγία είναι σημαντικό εργαλείο για το όλο οπλοστάσιο της πολιτικής ασύλου. Θέλουμε ένα ισόρροπο, δίκαιο, αποτελεσματικό σύστημα το οποίο μας ταυτόχρονα να μην κοστίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επομένω το θέμα οικονομικές επιπτώσεις για κάθε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάναμε έρευνα, ενδελεχή όταν υπευλήθησαν αυτέ οι προτάσεις οδηγιών σε σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για τι ε, μελέτες επιπτώσεων. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε στατιστικές πληροφορίες και σε δεδομένα που μας έδωσαν τα κράτη-μέλη όσον αφορά κάποια ερωτηματολόγια τα οποία εμείς τους απεστήλαμε. Μόνο ο λίγα κράτη-μέλη μας είπαν το πλήρες κόστος των διαδικασιών του ασύλου. Άλλοι μας υπέδειξαν κάποια στοιχεία, κυρίως όσον αφορά την δικαστική αρρωγή και κόστος του διερμηνίας. Ανάλογα με τις πληροφορίες λοιπόν προχωρήσαμε. Θέλουμε να συρρυκνώσουμε τα έξοδα. Θέλουμε η προσέγγιση μας να είναι ως εξής. Να μπορέσουμε να επενδύσουμε τους πόρους που έχουμε στα πιο πρώιμα στάδια της ε, διαδικασίας. Επομένως, στον πρώτο βαθμό αυτής της διαδικασίας, εάν επενδύσουμε, θεωρούμε ότι θα πετύχουμε αποτελεσματικότητα. Και νομίζω ότι ε, αυτά τα έξοδα θα αποσβεστούν από το ότι θα έχουμε λιγότερα έξοδα ή στους άλλους βαθμούς δικαιοδοσίας. Αυτή μας η προσέγγιση δικαιώθηκε από την έρευνα του Σόλιχαλ του Σεπτεμβρίου 2010 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιβεβαιώθηκε έτσι το ότι μια τέτοια μέθοδος που προσέχει τα πρώτα στάδια η νομικής ε, συμβουλής στα πρώτα στάδια με το να επιτρέπουμε τους νομικούς εκπροσώπους να συνοούνται με, τις, με αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις βελτιώνει την ποιότητα ή στην λήψη αποφάσεων σε πρώτο βαθμό. Και έτσι έχουμε γρηγορότερες αποφάσεις και περισσότερες θετικές αποφάσεις σε πρώτο βαθμό. Λιγότερες προσφυγές, εφέσεις, οτιδήποτε και λιγότερες επαναπροωθήσεις προς τη χώρα προώθησης. και τα εξόδα πρόνοιας, περίθαλψης, στέγασης και αυτά θα μειωθούν. Και κάποιες επιπλέον δαπάνες νομικής ε, προστασίας. Έχουμε επίσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία μελέτη όσον αφορά την κατανομή του βάρους μεταξύ των κρατών μελών που δέχονται τους ε, ετούντες άσυλο και Γι' αυτό θεωρούσαμε πάρα πολύ σημαντική πτυχή τον παράγοντα κόστος. Εμπειρικές, εμπειρικά στοιχεία επιβεβαίωσαν τις μελέτες και επίσης η μία μελέτη επιβεβαίωσε την άλλη. Άρα θα κάνουμε εμείς και άλλη μελέτη. Όμως, έχουμε τις επόμενες φάσεις των διαπραγματεύσεων όσον αφορά την οδηγία για τις διαδικασίες του ασύλου, οπότε και εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε στο πίγνιο της προσοχής μας την πτυχή, τον παράγοντα κόστος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Επίτροπε Φίλε, ευχαριστούμε για τα όσα μας εκθέσατε και τώρα περνάμε στις παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων θα έχουμε τους αγορητές των κοινοβουλευτικών ομάδων. Ξεκινάμε με τον αγορητή του ΕΛΚ, κύριο Μπουσούτιλ, ο οποίος θα έχει δύο λεπτά στη διάθεσή. Uh, λοιπόν, κοιτάξτε, σίγουρα έχει μπλοκαριστεί το θέμα του ασύλου, το πακέτο ασύλου. Είναι ατυχέ αυτό. Κακή κατάσταση, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να αποτελεματωθεί το ζήτημα. Για πολλούς λόγους έχουμε κολλήσει. Συγκεντρωθήκαν πρώτα απ' όλα σε νέες προτάσεις Όλοι ξέρουμε όμως ότι έχουμε υφιστάμενο νομοθεσία που προσπαθούν να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Αυτό δημιούργησε μια δυσαρέσκεια μεταξύ κρατών μέλων. Δεν θέλουν να προχωρήσουν με νέους νόμους όταν έχουν προβλήματα με τους ισχύοντες. Δεύτερον, οι νέες προτάσεις περιέχουν πολύ μεγαλύτερες υποχρεώσεις και βάρη. Και καμία φορά αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, κυρίως στο παρόν πλαίσιο. Και όπως αναφέρθηκε ήδη, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταχρήσεις, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί. Τρίτον, πράγματι υπάρχει έλλειψη μελέτης οικονομικής για να καθοριστεί το κόστος. Διαφωνώ μαζί σας κύριε Επίτροπε. Η μελέτη που διενεργήθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον μερισμό των βαρών δεν ε, αφορά μόνο το κόστος αυτών των προτάσεων. Ε, είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξετάσει τελικά τις οικονομικές συνέπειες των προτάσεών της. Μετά, δεν υπάρχει καμία πρόταση για νομικά, ένα νομικά δεσμευτικό μηχανισμό η κατανομή των βαρών. Και αυτό δημιουργεί δυσκολίες για κάποια κράτη-μέλη, αλλά και για το κοινοβούλιο μας. Τέλος, το Συμβούλιο εξακολουθεί να κολλησιεργεί όσον αφορά τις προτάσεις για την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου. Με τα χαράς άκουσα το Συμβούλιο να λέγει ότι η Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή και θα καταβάλει προσπάθειες για την εξέβρεση λύσεως όσον αφορά το θέμα του Δουβλίνου. Άρα δύσκολο το θέμα, δύσκολη η κατάσταση και πρέπει να ξεφύγουμε. Η ομάδα του ΕΛΚ είναι ανοιχτή θέλει να συνεργαστεί με το Συμβούλιο και πιο σημαντικό με άλλες ομάδες πολιτικές του Κοινοβουλίου για να καταλήξουμε σε αποδεκτό συμβιβασμό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Σεσίλια Δίξτρο από τους Φιλελεύθερους. Δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να ακολουθούν χρονοδιαγράμματα και έχουμε προθεσμία το 2012. Τότε πρέπει να είναι έτοιμο το κοινό σύστημα ασύλου προς χρήση. Έχω ελπίδες αλλά και ανησυχώ για αυτή την ημερομηνία. Θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα ή όχι. Υποτίθεται ότι θα έχουμε ένα κοινό σύστημα ε, για να γίνεται η έρευνα και να λαμβάνονται αποφάσεις για τις αιτήσει ασύλου και να αποφασίζουμε για το μέλλον των ανθρώπων. Υπάρχει παρόμοια κατάσταση. Θα, είναι, θα ισχύει παρόμοια κατάσταση όλα τα κρατήματα θα ισχύει το σύστημα. Σήμερα υπάρχουν τεράστιε διαφορέ. Δηλαδή η αντιμετώπιση των αιτήσεων διαφορετική, ποικίλη από κράτο μέλο σε κράτο μέλο. Και η έκθεση που ο Επίτροπο Φίλε μα ανέφερε ε, δείχνει ότι υπάρχουν τεράστιε διαφορέ μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Ξέρουμε επίση ότι μειώνεται το κόστο και μειώνεται το κόστο όταν βελτιωθεί η ποιότητα τη διαδικασία και λαμβάνονται σε πρώτο βαθμό οι αποφάσει. Θέλουμε να αλλάξουμε λοιπόν την οδηγία περί διαδικασιών και για μας θα είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο να ξέρουμε ποιο θα είναι το πραγματικό κόστος για το οποίο συζητούμε για τα κράτη-μέλη όταν μιλάμε για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου. Νομίζω με μια λεπτομερή ανάλυση των δαπανών θα αποφύγουμε σφάλματα. Και θα αποφύγουμε και σφάλματα που θα γίνονται εις βάρος των ετούντων. Ε, θα ήταν χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να μας δώσει πολύ λεπτομερέστερα στοιχεία, ανάλυση και να μας δείξει πώς μπορεί να μειωθεί το κόστος κατεργασίας, επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου. Και όπως είπε και ο αξιότιμος συνάδελφος κ. αυτό ίσως να είναι το κλειδί το κλειδί για να ξεφύγουμε από την αποτελμάτωση των συζητήσεων στο Συμβούλιο. Ελπίζω να είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Κρίμα που έχει κολλήσει το Συμβούλιο και πρέπει να βρούμε τώρα έναν τρόπο να ξεκλειδώσουμε την κατάσταση. Ακούσαμε τα όσα μα είπε ο Ούγγρος Πρωθυπουργό, που είναι επιφορτισμένο από την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και απευθύνω έκκληση στην Ουγγρική Προεδρία να συνεχίσει την έξοχη δουλειά που έκανε η Βελική Προεδρία. Θα ήταν πραγματικά κρίμα αν τελικά αυτή η διαδικασία κολλήσει τώρα. Ε, όλοι μαζί νομίζω θα μπορέσουμε να έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα σύλλου που θα έχει ένα ανθρώπινο πρόσωπο και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε το 2012. Συνεχίσουμε λοιπόν. Υπάρχει ακόμα ίχνος ελπίδας και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ρούι και από την Ενωτική Αριστερά. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι σε αυτές τις συζητήσεις ε, υπάρχει κάτι που, συμπερι, ε, που εμπεριέχεται. Δηλαδή, να μην είναι ακριβό, λέει το, η ανθρωπιστική προσέγγιση. Όμως αυτό όμως ε, υπάρχει και, το ότι αν είναι δαπανηρό θα πρέπει να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει για την ανθρωπιστική προσέγγιση. Δηλαδή, η ανθρωπιστική προσέγγιση είναι μια πιο ε, φθηνή προσέγγιση. Και σε σχέση με το σώμα ε, το νομοθετικό στην Βρετανία που είχα παραστεί, είναι το πιο δαπανηρό πανηρό είναι η καθυστέρηση και ε, τα προβλήματα που δημιουργούνται για τις οικογένειες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι έχουμε το πρόβλημα το διοικητικό, διοικητικό κόστος για εκείνους που ε, ετούνται άσυλο και για άλλους που για οποιονδήποτε λόγο έχουν τύχη αρνητικής απάντησης. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα. Αν είναι δυνατόν να υπάρχει μια ε, ανθρωπιστική προσέγγιση που θα είναι και λιγότερο δαπανηρή, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Και θα πρέπει να δούμε ότι ότι αν υπάρχει εδώ πρόβλημα δεν είναι μόνο το ότι υπάρχει θέμα δαπανών από τα κράτη-μέλη αλλά επειδή είναι μερική η υλοποίηση αυτών των διατάξεων και είναι η καταστολή η οποία υιοθετείται. Εδώ για τους ετούντες άσυλο και για τις ε, εθνικές διοικήσεις πρέπει να δούμε σε τελευταία ανάλυση τι μπορεί να δει. Θα πρέπει να μας δώσει το Συμβούλιο τα στοιχεία ε, απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις και να υπάρχει μια συνεκτική δράση και τοποθέτηση για να είμαστε αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Και στη συνέχεια θα περάσουμε στον επόμενο αγορητή, Gerard Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Αυτή η συζήτηση απορρέει από την ανάγκη για να υλοποιηθεί το σύστημα το οποίο προβλέπει στην της Λισαβόνα στα κράτη-μέλη χάνουν ακόμη περισσότερο έλεγχο της μοίρα τους ή αν πρέπει να πληρώσουν ε, ένα κόστος το οποίο ακόμα είναι ανυπολόγιστο. Ε, το ήδη το σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα χάος. Έχουμε χιλιάδες υποθέσεων που εκκρεμούν και ε, πάρα πολλοί επίσης ε, έχουν εισέλθει στη χώρα παρανόμως και αυτό δεν βοηθάει τίποτα τη μετανάστευση, τη νόμιμη. Καταλαβαίνω ότι πάνε χαμένα τα λόγια γιατί οι περισσότεροι από εσά δεν νοιάζονται για το κατά πόσον θα περισσωθούν οι δημοκρατικές δυνάμεις του, του, του, κράτους έθνους. Οι περισσότεροι βρισκόταν σε αυτή την φαντασίωση της ε, αενά ολοκλήρωσης ε, που είναι κάτι σαν τους πίνακες του Ιερώνιμου Μπός, όμως ο λαός στη Βρετανία πρόκειται να αναζητήσουν τους υπεύθυνους, αυτούς οι οποίοι επρόδωσαν τους πολιτικάντιδες, οι οποίοι δεν τους έδωσαν την ε, ευκαιρία να, να κάνουν δημοψήφισμα για τον Εμένο Βασίλειο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ομπερμάγερ στη συνέχεια. Παρακαλώ ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μέχρι το 2012 το δικαίωμα για το άσυλο θα ενιοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις ε, ταχύες απελάσεις ε, σε σχέση με ε, περιοχές διαμετακόμισης θα είναι εφικτές τέτοιες δράσεις. Όμως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις ε, διεργασίες στα αεροδρόμια λέει ότι πρέπει να συνεχίσει να είναι δυνατόν ε, οι ετούντες άσυλο στα σύνορα να μην γίνονται δεκτοί και να επιστρέφουν. Γνωρίζουμε τη συζήτηση. Τι σημαίνει ασφαλής χώρα προέλευσης και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για αυτό το θέμα στην Ευρώπη. Προβλέπετε επίσης ότι θα δίνονται δικαιώματα σε συγγενείς όπως ε, για παράδειγμα σε σχέση με τους ε, ε, γονείς ή τους συζύγους των ετούντων άσυλο. Θα πρέπει να δούμε σε βάθος αυτές τις προτάσεις οι διαδικαστικές διεργασίες και το κόστος πρέπει να μας κάνει να δούμε ότι θα υπάρξει μικρότερη γραφειοκρατική επιβάρηση και μικρότερο κόστος και δυστυχώς υπάρχει και η προοπτική να υπάρξει ολόκληρο κύμα τέτοιων ανθρώπων που θα στην Ευρώπη και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ και ολοκληρώσαμε τώρα πλέον με αυτόν τον τρόπο τον επίσημο κατάλογο εκείνων που ε, θα μπορούσαν να παρέμβουν από πλευρά των κοινοβουλευτικών ομάδων. Περνάμε τώρα στις περαιτέρω παρεμβάσεις ατομικά των Ευρωβουλευτών. Ο κύριος Γιακολίνο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σίγουρα αυτή η οδηγία για τις διαδικασίες έχει ιδιαίτερη σημασία το καθεστώς του πρόσφυγα πρέπει ε, να εξετάζεται με αυστηρότητα και επιβάλλει λοιπόν η διαδικασία της αναγνωρίσης του καθεστώτος του πρόσφυγα να είναι γρήγορη και ευέλικτη και αυτό ειλικρινά δεν είναι κάτι που συμβαίνει. Ε, στο Συμβούλιο έχει κολλήσει το πακέτο για το άσυλο που θα πρέπει να καθορίσει ένα νέο πιο σύγχρονο πλαίσιο αναφοράς και εντωμεταξύ ε, δείχνει ότι υπάρχουν διαφορετικοί προστατευτισμοί από τα κράτη-μέλη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ασύλου. Όσον αφορά τις, σε σχέση με του νόμου που ήδη εφαρμόζονται, στρέφομαι προ τον Επίτροπο που είναι εδώ. Δεν μπορούμε να επικαλούμεθα την κρίση για να μειώσουμε τη χρηματοδότηση που είναι αναγκαία όσον αφορά τη διαδικασία που είναι σημαντική ανάμεσα στα άλλα επιχειρήματα που δεν θεωρώ ότι όλα τα επιχειρήματα είναι πιστικά έναντι μια διαδικασίας ε, που έχει κολλήσει. για να μην κολλήσουμε εκεί, θα πρέπει να, θα, για να κολλήσει εκεί υπάρχουν ε, διάφοροι λόγοι πολιτικοί, θρησκευτικοί κλπ. Ε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που ζητούν άσυλο έχουν δικαίωμα υποδοχή στα κράτη-μέλη. Και είναι αναγκαίο να αρνηθούμε το δικαίωμα υποδοχή όταν κάποιο ισχυρίζεται ότι είναι ε, πρόσφυγα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Πράγματι το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη έχει ε, θεσπίσει αυτή την αρχή τα τελευταία δύο χρόνια 250.000 ε, εξετάστηκαν και είναι πολύ σημαντικός αριθμός αν και έχει μειωθεί με το έτος αναφοράς. Ε, χρειάζεται διερμηνία, παροχή συμβουλών, χρειάζεται μείωση των δαπανών και χρειάζεται ισορροπημένη κατανομή των βαρών. Χρειάζεται πιθανότατα μια καλύτερη λειτουργία όσον αφορά των διαφόρων υπηρεσιών υποστήριξη, ε, όπω είναι αυτό στη Μάλτα, χρειάζεται με Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματικά θα πρέπει να κάνει ένα βήμα μπροστά αποφασιστικό, ούτω ώστε να εγγυάται τα δικαιώματα στου πρόσφυγε και ταυτόχρονα όμω να εισαγάγει στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, ε, να καθορίζεται ποιος έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μωράης στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο. Δύο λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπε και η συνάδελφος Γκυγιόμ, είναι πάρα πολύ κρίσιμη η συγκυρία για την εξέλιξη της πολιτικής ασύλου. Σε κάποιες με τις διαδρομής τα πήγαμε καλά με τη Βελική Προεδρία και τη Διεθνή Προστασία, όμως αυτά όλα είναι παρελκόμενα για το όλο πακέτο τη δέσμη των μέτρων, γιατί θα πρέπει τώρα να δούμε τι γίνεται ακριβώ με τι πονδυλικέ στήλε τη υπόθεση. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε βήματα προόδου, να δούμε τι θα γίνει με την καταλητική προθεσμία του 2012, που πρέπει να έχουμε φτιάξει το σύστημα και έχουμε τι επικρίσει των κρατών μελών σε σχέση με αυτέ τι νέε διαδικασίε τη αναθεώρηση του συστήματο. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το, με το βάρο των δαπανών. Όμω υπάρχουν εδώ πέρα διάφορα ε, στοιχεία, είπατε και για, το, για τη μερίδη του Σόλιχαλ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και εδώ πέρα έχουμε στοιχεία πολλά που οδηγούν και κατατείνουν στο ότι το front loading, δηλαδή το να, το να τα δώσουμε όλα στις πρώτες φάσεις οδηγεί σε, σε, σε επιτυχία. επομένω, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Αν θέλουν τα κράτη-μέλη να υποστήριξουν τα επιχειρηματικά, να δώσουν περισσότερα στοιχεία. επομένω το θέμα δεν είναι τώρα μόνο τα κόστη το, όλο το προτσές που χρειάζεται μία εναρμόνιση και να πάει ο πύχης στον στάνταρ ε, πιο ψηλά και να δούμε που χρειάζεται να διορίσει και το νομικό πλαίσιο, το νομικό καθεστώς. Θα μας όμως μήνες να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι χρειάζεται και να δούμε τι θα πει και το Συμβούλιο. επομένω εμείς ήμασταν αποφασιστικοί και θέλουμε να μην απονευρωθεί η πρόταση της Κομισιόν από το Συμβούλιο το δικαίωμα σε νομική αρρωγή επίσης, να κατοχυρωθεί, προσοχή για τις επιταχυμένες διαδικασίες και να καταλήξουμε σε αποτελεσματικό σύστημα. Έτσι θα πετύχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα. Στόχος του Κοινοβουλίου θυμάμαι ότι είναι αυτός από το, το 1999 στο Τάμπερε, το Συμβούλιο τα είχε πει. Στη Χάγη τα ξαναείπανε και στη Στοκχόλμη. Άρα να σταθερήσουμε την ιστορία και επομένως απόκειτο στο Συμβούλιο τώρα να απεμπλέξει την κατάσταση. Μέσα σε συνεργασία με την Προεδρία προσπαθήσουμε να συνεχιστεί η φόρα που πήρε το θέμα από τη Βελική Προεδρία. Καλά, δεν συμφωνούμε όλοι. Ας ελπίσουμε όμως όλοι ότι με την Προεδρία την τωρινή θα δούμε κάποια πρόοδο. Μάλιστα, σωστό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντίεστε Μέρα παρακαλώ. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ και για την κοινή πολιτική, για το θέματα, για τα θέματα ασύλου. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Σεπτεμβρίου τονίζει τα πολλά πολυάριθμα εμπόδια που αντιμετωπίζουν το κράτη-μέλη όταν έχετε στιγμή να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας αυτής το δικαίωμα των ετούντων άσυλο που πρέπει να έχουν σύνδρομη ε, αφορά διαφορετικά επίπεδα Πολλά κράτη αναφέρονται στις ε, απαιτήσεις αυτής της οδηγίας ε, σε σχέση με τη συνδρομή, αλλά αναγνωρίζουν και το, τη διαδικασία ε, ε, σύνταξης της αίτησης ασύλου και ε, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Και εδώ θα έχουμε και το θέμα και της δωρεάν συνδρομής. Στις, στην πλειοψηφία έχουμε διαφορετικές δυνάμεις που επενεργούν, ενώ έχουμε και το θέμα της αυτόματης Άσεις ε, όταν έχουμε αρνητική απάντηση δημιουργεί και αυτή προβλήματα καθώς εφαρμόζεται ή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε έξι κράτη-μέλη. Όλες αυτές οι διαφορές τονίζουν ότι ο μηχανισμός που αφορά αυτή την οδηγία θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Και για αυτή την αναθεώρηση συμπίπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάγκη του να επικεντρωθούμε στην αρχική φάση της εφαρμογής, όντας περισσότερο αποτελεσματική στη στιγμή που διαφοροποιούμε ποια άτομα έχουν ή όχι δικαίωμα δικαίωμα για προστασία που θα τους χορηγηθεί. Και αυτού, αυτό το μέτρο θα συνεισφέρει σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής να υπάρξουν εξοικονομήσεις δαπανών και να παραμείνουμε σε ένα χαμηλότερο κόστος. Όποιο, όμως πρέπει να δούμε εξειδικευμένα ποια θα είναι τα κόστη της συνδρομής και της διερμηνίας πρωτοβάθμια και το κόστος το οποίο θα επιβαρύνει, θα επιβαρύνει τα κράτη-μέλη. Για αυτούς όλους τους λόγους είναι αναγκαίο να ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πραγματικά κόστη τα οποία θα συνεπάγεται η πρόταση αυτή που ε, υποβάλλεται. Και δεν θεωρώ ότι είναι αποδεκτό με την αρνητική τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη αυτή η θέση και πρέπει να επανεξεταστεί ή να διαφοροποιηθεί. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρόμερο Λόπες θα λάβει τώρα τον λόγο. Δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Υφυπουργέ, σας καλωσορίζουμε στο Ευρωκοινοβούλιο που ήταν και δικό σας, δικό σας χώρος και Θεωρούμε ότι ακόμα και αν αυτό το θέμα δεν ήταν ε, εν σας ε, δείχνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα ασύλου. Θέμα το οποίο προωθήθηκε από την Βελγική Προεδρία και την χάνει και προώθησης από την Ουγγρική Προεδρία και θέλουμε να αναφέρουμε ότι αληθεύει ότι αν μπορέσει να προωθήσει αυτά τα θέματα η Προεδρία και να έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα στοιχεία που χρειάζονται. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες ε, που συνεπάγονται σε σχέση με την πρόταση αυτή και υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν είναι πρόθυμα να διαθέσουν τέτοια στοιχεία, δεν μπορούν να τα διαθέσουν και δεν έχουν γίνει εκτιμήσεις ε, για... Ε, και δεν έχουν ακολουθηθεί σωστές διαδικασίες. Όμως αυτά τα κράτη κράτη-μέλη ίσως ε, μπορεί να θεωρήσουν ότι αυτή η αναθεώρηση αυτού του πλαισίου πρωτοβάθμια θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του κόστους ε, και σε σχέση με τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση κιόλα ε, λόγω αυτού του φαινομένου του, των ετούντων άσυλο. Και έχουμε εδώ διαφορές διαδικαστικές. Κάποια κράτη επιβαρύνονται περισσότερο από άλλα σε σχέση με τους ετούντες άσυλο. Με αυτού του είδους την πρόταση θα, θα εξοικονομούσαμε πολλές ε, δαπάνες ε, και το κόστος για το άσυλο θα ήταν μικρότερο. Θα ενιοποιούσαμε τις διαδικασίες και θα διευκολύναμε τις διεργασίες, διότι κάνουμε λόγο όχι μόνο για το κόστος για αυτές τις διεργασίες, αλλά κυρίως ε, στην ουσία αυτό το, για το οποίο συζητάμε είναι το κόστος το οποίο συνεπάγεται το να μην έχουμε ένα κοινό ενιαίο σύστημα για το άσυλο. Και βλέπουμε τι συμβαίνει στα εξωτερικά σύνορα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης με άτομα τα οποία Ισραήλ θέλουν να ε, καταλήξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προέρχονται από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ και από χώρες που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Πρέπει να υπάρχουν τα αναγκαία εχέγγυα ώστε να αντιμετωπίζονται σωστά αυτοί οι άνθρωποι να μην καταλήγουν σε κέντρα υποδοχής ε, επί μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ε, κανένα είδος ε, συνδρομής και πρέπει να δούμε ποιο είδος καθεστώτος θα τους δίνεται ή όχι και βλέπουμε ότι το κόστος το οποίο συνεπάγεται αυτό, αυτή η κατάσταση με το να παραμένουν αυτά τα άτομα σε τέτοιους καταβλισμούς ή τέτοια στρατόπεδα που επειδή δεν είχαν τα χρήματα να ε, μπορέσουν να μεταβούν διαφορετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε ότι αυτές οι τραγωδίες ε, πρέπει να αποφευθούν ή να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σαν τέτοια δεν και ο κατάλογο ε, των ομιλητών δηλαδή. Και τώρα όμω έχει το λόγο ο κύριο του... Όχι ο κύριος Παπα-Νικολάου, αλλά ο κύριος Κοέλιο, ο οποίος θα έχει δύο λεπτά στη διάθεσή του για την παρέμβασή του. Ο κύριος Κοέλιο, λοιπόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινάω, Πρόεδρε, συγχαίροντας τους συντάκτες αυτής της ερώτησης και την κυρία Μόνικα Χολμάιερ ευθυγραμμίζονται αυτά με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δίας Δεμέρα. Βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα από τα πέντε μέσα που έχουμε για την αντιμετώπιση των θεμάτων ασύλου, για τι ελάχιστε προδιαγραφέ που θα εφαρμόζονται διαδικαστικά για του ετούντε άσυλο. Όμω στην έκθεση που μα υπέβαλε πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζεται το γεγονό ότι τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν διαφορετικέ πρακτικέ και ότι υπάρχουν διαφορέ, πολύ σημαντικέ διαδικαστικά σε σχέση με το πώ αντιμετωπίζονται αυτά τα άτομα που ετούνται άσυλο και έχουμε σημαντικότερε διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών. Έχουμε λοιπόν επιταχυμένε συνοπτικέ δικαστικές διαδικασίες καθώς επίσης και την χορήγηση ε, σύνδρομης ή πραγματική αποτελεσματική βοήθεια. Να το πούμε ξεκάθαρα. Κράτη-μέλη με μη σωστό τρόπο ή ελλειπή τρόπο υλοποίησαν αυτή την οδηγία και άλλα κράτη-μέλη απλά την εφαρμόσουν πολύ χαλαρά και καθόλου αυστηρά. Λοιπόν, διήνθατερον, ή θα πάψουμε να έχουμε αυτή την κατάσταση ή θα πρέπει να αρθεί αυτή η διαφορά και να καταλήξουμε σε ένα κοινό σύστημα. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, να υπάρξουν βελτιώσεις, βελτιώσεις που είναι αναγκαίες και να έχουμε τη διαδικασία front loading, να ξεκινήσουμε σε πρώιμο στάδιο. Είναι αναγκαία λοιπόν η παρέμβαση της Επιτροπής, είναι αναγκαίο να ταυτοποιήσουμε πού μπορούμε να βελτιώσουμε κάτι και για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διαφορές. Να δούμε ότι χρειάζεται συνεργασία των κρατών μελών σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Συμπεριλαμβάνοντας, αλλά όχι μόνο βέβαια, το θέμα του κόστους. Και ιδιαίτερα θα πρέπει από πλευρά ε, της Ευρώπης και τα κράτη-μέλη να καλύψουν αυτόν τον στόχο, να πετύχουν αυτόν τον στόχο. Ο στόχος μας πρέπει να συνεχίσει να είναι ο ίδιος. Το 2012 με άλλα λόγια να καταλήξουμε σε ένα κοινό σύστημα για το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα γίνει πραγματικό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, Σα ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητέ συνάδελφε, και τώρα τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό: ο κύριο παπα Παπα-Νικολάου παρακαλώ. 1,5 λεπτό παρακαλώ κύριε Παπα-Νικολάου. Πρόεδρε, ξέρω ότι μοιάζουμε με τον κύριο Κοέλιο, γι' αυτό και μας μπερδέψατε προηγουμένω. Ε, και θα μιλήσω συγκεκριμένα. Σήμερα σήμερα μόλις η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της να σταματήσει να επαναπροωθεί πρόσφυγες στην ελλάδα για τους επόμενους δώδεκα μήνες και ανάλογες αποφάσεις έχουν ληφθεί από τη σουηδία τη μεγάλη βρετανία την ισλανδία και την νορβηγία. ωστόσο μόλις πριν από λίγους μήνες τον περασμένο νοέμβριο το συμβούλιο των υπουργών δικαιοσύνης δεν δέχτηκε τη συμπερίληψη ενός μηχανισμού αναστολής μεταφοράς των ετούντων άσυλο στον αναθεωρημένο κανονισμό δουβλίνο 2, όπως είχε προτείνει η επιτροπή από το 2008 και θεώρησε το συμβούλιο πριν από δύο μόλις μήνες ότι το δουβλίνο 2 έχει καλώς και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. την ίδια στιγμή επιθυμούμε και καλώς κάνουμε και αυτό οφείλουμε να πράξουμε με την οδηγία που σήμερα συζητούμε την παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης προς τους αιτούντες άσυλο στον πρώτο βαθμό εξέτασης του αιτήματός τους. γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι και αναφέρθηκε προηγουμένως αυτό και από την κυρία χολμάιερ ότι αυτές τι διαδικασίες πολλές φορές τις καταχρώνται οι αιτούντες προκειμένου ενώ δεν το δικαιούνται να παρατείνουν όσο μπορούν με νομικά τερτύπια αν θέλετε τη διαμονή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος και όλα αυτά χωρίς να έχουμε σαφή αξιολόγηση για το κόστος ενός τέτοιου μέτρου και το κατά πόσο αυτό θα υπονομεύσει στη συνέχεια την υλοποίησή του. και διαρωτώ με τελικά αγαπητοί συνάδελφοι με τέτοιες αντιφατικές αποφάσεις πώς θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ένα βιώσιμο κοινό σύστημα ασύλου ως το 2012 όταν εμείς οι ίδιοι άλλα αποφασίζουμε άλλα προτείνουμε και τελικά άλλες ενέργειες κάνουμε και άλλα αποτελέσματα έχουμε στην πράξη είναι αυτό για λόγους αδυναμίας είναι λόγω του ελλείμματος αλληλεγγύης ή κάτι άλλο που ενδεχομένως μπορεί να μας διαφωτίσει το συμβούλιο και η επιτροπή. σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Τρεις έχουν ζητήσει να παρέμβουν και οι τρεις θα μπορέσουν να παρέμβουν. Λοιπόν, ο κύριος Αλώνε πρώτος. Ένα λεπτό παρακαλώ κύριε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ δεν θα ήθελα να θέσω λάθος τόνο στη συζήτηση. Είμαι πεπισμένος ότι ο συσχετισμός και από σημειολογική έποψη και όσον αφορά την εξοικονόμηση και σε σχέση με το δικαίωμα χορηγήσεως ασύλου ε, έχουν σχετισμό αρνητικό. Να εξηγηθώ τι θέλω να πω. Δηλαδή, πιστεύω το πρόβλημα το πραγματικό είναι η εναρμόνιση και όχι το διοικητικό κόστος. Δεν είναι ιδεολογικό πρόβλημα, αλλά κυρίως πολιτισμικό. Δυστυχώς υπάρχουν πολιτισμικές προσεγγίσεις. Όχι ιδεολογικές. Αυτό πρέπει να δούμε. Οι πιο κρεθυμένες χώρες είναι οι μεσογειακές. Έχουν πολιτισμό υποδοχής πολύ πιο ισχυρό από άλλες χώρες. Διόχουμε έχουν σχέση πολύ πολύ πολύ πιο στενή με αυτό το πρόβλημα. Ενώ στην Ιταλία αυξήθηκε αυτή η δαπάνη. Αυξήθηκε, φτάσαμε στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Σε άλλες χώρες θέλουν να μειώσουν το κόστος. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πρέπει να προσέξουμε να δώσουμε ένα πέμπτο αυτών των δαπανών όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα για τα προβλήματα των αναπήρων. Γιατί πολύ συχνά ο πολιτικός πρόσφυγας είναι και ένας άνθρωπος που έχει αναπηρία. Διότι υπέστη βασανιστήρια. Όπως θα πρέπει να συζητήσουμε επίσης και για προστασία των ανθρώπων που προστατεύονται. Είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, η προστασία κάποιων ατόμων που πρέπει... Για αυτή την προστασία δεν άκουσα τίποτα να λέγεται. Στην Ευρώπη των ελευθεριών στην Ευρώπη της προστασίας των δικαιωμάτων. Και διακόπτε το μικρόφωνο του ομιλητού. Ναι, όμως ήδη δύο λεπτά σχεδόν μιλούσατε αντί ενός λεπτού. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Ευρωβουλευτά. Και τώρα θα ακούσουμε την Ελένα Μπασέσκου. Έχετε ένα λεπτό κυρία Παρακολουθή. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. αυτή, αυτή η οδηγία που πρέπει να αλλάξει όσον αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές και ρήτρες για τη χωρίση ασύλου πρέπει να διαμορφωθεί πιο αποτελεσματικά και πρέπει να υπάρξει απλούστευση και ε, ενιοποίηση των διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διατάξεις και ρήτρες πρέπει να προσανατολίζονται στις βέλτιστες πρακτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζουν έτσι αυτές τις περιπτώσεις. Όμως έχουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα σε σχέση με τα εθνικά συστήματα. Έχουμε μεγάλες διακοιμάνσεις ε, και ε, διαφορές. Αυτό οδηγεί σε μεγάλα προβλήματα διοικητικά που το δυνατόν ταχύτερο θα έπρεπε να επιληθούν από μια κοινή προσέγγιση. Ζητώ λοιπόν από το Συμβούλιο το δυνατόν ευρύτερες πληροφορίες να συλλέξει από τα κράτη-μέλη, πληροφορίες που θα δοθούν ώστε να ξεκινήσουν οι νέες ε, διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσει, ώστε έγκαιρα, εμπρόθεσμα να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Σα Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Ευρωβουλευτά. Τελευταίος εξίσου σημαντικό σε σχέση με την παρέμβαση η κυρία Βρονμάη. Είναι μία από τις συντάκτριες και έχει τον λόγο πάλι. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που μου δίνετε τον λόγο σύντομα. Έχω μια μεγάλη παράκληση προς εμάς κύριε Επίτροπε Φιούλε. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι οι, οι λάθος υποθέσεις και οι υπολογισμοί οδηγούν σε λάθος κόστος. Και εδώ έχουμε και θέματα όσον αφορά και τις χορηγήσεις θεωρήσεων διαβατηρίων σε σχέση με την Σερβία, Μακεδονία, λέει ομιλήτρια. Υπάρχουν μεγάλες προσπάθειες κατάχρησης ε, αυτού, αυτής της δυνατότητας να προσέχουν σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ξεκινά κανείς από εσφαλμένες υποθέσεις ε, ή επιχειρήματα και λέει ότι ε, μια τέτοια διαδικασία θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση κόστους τότε υποθέτει κανείς ότι σε όλα τα κράτη-μέλη πρωτοβάθμια ισχύει μια αρνητική κατάσταση. Δεν ισχύει όμως αυτό. Αν δούμε το τι σημαίνει και ποια θα είναι η επίπτωση για την αύξηση του κόστους, αύξηση των, ε, και αναβάθμιση των ποιοτικών προδιαγραφών, είμαι πρόθυμη να συζητήσω στην πραγματικότητα τι θα δημιουργηθεί. Μεγαλύτερο κόστος κόστος και πρέπει εδώ να δούμε και τις ε, ενστάσεις και επιφυλάξεις που έχουν τα κράτη διότι υπάρχουν αυτές οι τοποθετήσεις και πρέπει να λυθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε. Και έτσι τώρα σχεδόν φτάσαμε στο τέλος ε, των εργασιών μας. Ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Επίτροπο Φιούλε να τοποθετηθεί. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ισότιμοι κύριοι βουλευτές, άκουσα με μεγάλη προσοχή τις απόψεις των μελών του Κοινοβουλίου. Η διαδικασία αυτή για το άσυλο είναι πολύ σημαντική για το σύστημα που θα πρέπει να έχουμε συγκροτήσει μέχρι τέλους 2012. Χαιρετίζουμε την δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προχωρήσει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις για την σχετική οδηγία και όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο, η Επιτροπή επίσης θεωρεί πάρα πολύ θετικό το πόσο δεσμεύονται τα κράτη-μέλη να υπάρξει μια συνεννόηση ανοιχτή και επικοδομητική και πάρα πολλές από τις προτάσεις τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τις εκπαιρεώσουμε και γι' αυτό και εμείς πρόκειται να διατροποποιήσουμε την πρότασή μας πριν την αρχή της Πολωνικής Προεδρίας. Ο απότερος στόχος μας είναι να σημειωθεί πρόοδος προς μια κοινή διαδικασία και να διευκολύνουμε αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων της διαδικασίας. Οπότε θα πρέπει βέβαια και με την τροβημένη πρόταση να εξασφαλίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και να υπάρχει λήψη αποφάσεων σε υψηλή απόφαση σε πρώτο βαθμό. Αυτό θα μας οδηγήσει σε συνέπεια των αποφάσεων και επομένως θα έχουμε και ζερίγνωση των εξόδων. Στην τροπημένη πρόταση η Επιτροπή θα προσπαθήσει να πλουστεύσει κάποιες διατάξεις και έτσι να πιο εύκολη εφαρμογή τους θα συνεχίσουμε να πασχίζουμε για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά το, την οικονομική πτυχή, καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι το θέμα κόστος για την πρόταση αυτή. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε το βάρος σε αυτή την πτυχή και στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Εν κατακλείδη θέλω να σας τονίσω ότι η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της επεξεργασίας της τροπεμένης πρότασης. Θα συνεχιστεί η συνεργασία μας με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. στα πλαίσια της δουλειάς μας για το Γενικό Ενέδες για το Άσυλο. Πρόεδρος. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και τώρα τελευταία αλλά πάρα πολύ σημαντική κυρία Ενικό Γκέρι που είναι η αρμοδία Υπουργός. Με την οποία κληρώνει το κατάλογο των αγορητών. Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και σας ευχαριστώ επίσης για το γεγονός ότι πραγματικά συζητήσαμε και μπορέσαμε να συζητήσουμε για πολύ συγκεκριμένα εξειδικευμένα θέματα. Είμαι σίγουρη ότι με τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα σημειωθεί πρόοδος και θα είναι αυτή αυτά όλα θα ληφθούν υπόψη και είναι σημαντικό αυτό. Χρειάζονται ελάχιστε προδιαγραφέ και ρήτρε. Είναι απόλυτα σαφέ αυτό. Πρέπει να ε, πάψουν να υπάρχουν ε, καταχρήσεις πρέπει να ε, προλάβουμε τις καταχρήσεις την κατάχρηση και είναι όλα αυτά προβλήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν από κοινού και θα τα ρυθμίσουμε μια σκέψη θα ήθελα εν τέλει να εκφράσω με υπερηφάνεια βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα. Μια κοινότητα όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι σεβαστή. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι μια από τις σημαντικότερες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το θέμα, για τα θέματα ασύλου, πρόκειται ακριβώς για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο αυτό σε αυτόν τον προσανατολισμό. Η, Ευρωπαϊκή, η Ουγγρική Προεδρία θέλει τον άνθρωπο να τον θέτει στο επίκεντρο σε όλους τους τομείς πολιτικών προηγούμενα προαναφέρθηκε ότι η σημερινή κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει τέτοια μορφή που πρέπει με πραγματογνωμοσύνη και νυφάλια να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Πρέπει όμως να δούμε και τη συναισθηματικά φορτισμένη πλευρά που είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Για παράδειγμα για τους Ρωμά, τους Τσιγκάνους. Πρέπει να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δρά όχι μόνο ορθολογιστικά με τον νορθό λόγο αλλά και συναισθηματικά ευχαριστώ και θέλω να πω ότι έχουμε και την πράσινη βίβλο είναι γνωστό αυτό, είναι διαθέσιμη σε όλους μπορεί κανείς να διαβάσει σε σχέση με αυτήν ποιες είναι οι προτεραιότητες των Υπουργών Εσωτερικών σε αυτή την προοπτική και ήδη και σήμερα το πρωί το προανέφερα στις ε, παρεμβάσεις που έκανα πραγματικά με όλους επιθυμούμε να συνεργαστούμε και θα συνεργαστούμε με όλους. Θέλουμε το δυνατόν γοργότερα στο Συμβούλιο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, ώστε με αυτόν τον τρόπο εσείς στη συνέχεια να μπορέσετε να εκφράσετε τη γνώμη σας και να πείτε ότι ορίστε, πραγματικά η Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου ενδιαφέρθηκε, με για αυτό το θέμα με θετικό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Υφυπουργέ, λέει ο Πρόεδρος. Και έτσι μπορώ να, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε απόλυτη, απόλυτα πλήρη εμπιστοσύνη στην Ουγγρική Προεδρία